Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Πρώτος ομιλητής είναι ο Επίτροπος Ντεχίχτ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ καθίστε, σας δίνω λίγο χρόνο να τακτοποιηθείτε. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, μετά από πέντε χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων, οι επικεφαλείς των διαπραγματευτικών ομάδων κατέληξαν και έχουμε ένα κείμενο συνολικό οικονομικής ε, και εμπορικής συμφωνίας Ένωσης Καναδά. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ έλαβε αμέσω το κείμενο το οποίο θα δημοσιευθεί συντόμω. Ο Καναδά είναι το πρώτο κράτο G8 με το οποίο έχουμε σφαιρικό κείμενο συμφωνία εμπορίου. Έχει ζωτική σημασία για την αξιοπιστία του εμπορικού μα θεματολογίου διότι επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλέ συμφωνίε με ανεπτυγμένε οικονομίε που έχουν τη δική του προσέγγιση και το δικό του ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό Υπήρχαν βέβαια δύσκολες φάσεις διαπραγμάτευση. Η συμφωνία είναι επίσης πολύ πολύτιμη αυτή εξ αυτή. Δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας. Ο Καναδάς είναι αρκετά μεγάλη αγορά για μας και <clears throat> οι δικές μας εταιρείε θα έχουν την ίδια και καλύτερη αντιμετώπιση από ότι οι επιχειρήσει των ΗΠΑ. Αυτό θα μας βοηθήσει για περισσότερη ανάπτυξη και θέσει εργασία στην Ευρώπη δεδομένων και των ανησυχιών που έχουμε αυτή τη στιγμή ο Καναδάς είναι σημαντικός μας εταίρος πολιτικά και σύμμαχος. Είναι επίσης σημαντικός προορισμός επενδύσεων και ο ίδιος ο Καναδάς επενδύει μαζικά στην Ευρώπη, δημιουργεί ανάπτυξη και απασχόληση. Έχει επίσης ίδιους πόρους και πρώτες ύλες. Μέσω λοιπόν αυτής της συμφωνίας ΣΥΤΑ και οι δύο πλευρές με πολύ λίγες εξαιρέσεις θα καταργήσουν όλους τους Τελωνιακού δασμού για μερικά πολύ ευαίσθητα γεωρικά προϊόντα θα παραμείνει προστασία. Επίσης θα ανοίξει η αγορά επενδύσεων και υπηρεσιών και έχουμε καλύτερη θέση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε που έχει την αυτά και όλες μας οι κυβερνήσεις θα έχουν δυνατότητα να παρέχουν και να επιδοτούν δημόσιε υπηρεσίε. Επίση θα έχουμε μεγάλη πρόσβαση στι δημόσιε προμήθειε. Μέσω του ΣΥΤΑ έχουμε μεγάλη πρόσβαση σε αυτέ τι αγορέ δημοσίων προμηθειών του Καναδά σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση. Η συμφωνία δημιουργεί νέε προδιαγραφέ για διαδικασία διαιτησία σε περίπτωση διαφωνιών για επενδύσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίε για αυτή τη συμφωνία και θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω όλε τι ανησυχίε που έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα. Θέλω να τονίσω επίση και το αποτέλεσμα για τα προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης. Έχουμε ένα αναλυτικό σύστημα προστασίας στον Καναδά για τα προϊόντα μας, ε, τα γεωργικά υψηλού επίπεδου Παρμιτζάνο Ρεζάνο, Σφαρσβάλτερ Σίνκεν, Μπλοντοβέρνιε και 142 άλλα προϊόντα που θα προστατευτούν πλήρως. Είναι ένα από τα τμήματα που καταδεικνύει σαφώς ότι η ΣΥΤΑ μπορεί να ωφελήσει και τις μικρομεσαίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σχέσεις μας στον εμπορικό και επενδυτικό τομέα βεβαίως δεν θα πρέπει να θίξουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές προδιαγραφές. Έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Έχουμε πολύ υψηλού επίπεδου προδιαγραφές. Υψηλότερες από ό,τι είχε ποτέ ο Καναδάς. Τα επόμενα βήματα ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο Καναδός πρωθυπουργός Χάμπαρ Προτίθεται να αναγγείλουν δημόσια την κατάληξη των δραματεύσεων στην Άζη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά τον, στην Όταουα στις 26 Σεπτεμβρίου και κατόπιν οι δύο πλευρές θα υποβάλουν τα κείμενα αυτά στις αντίστοιχες νομοθετικές αρχές για επαλήθευση και επικύρωση. Για την Ένωση αυτό σημαίνει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Επειδή ε, ε, ο νομικός έλεγχος και οι μεταφράσεις παίρνουν χρόνο, υποθέτω ότι η υπογραφή στο Κοινοβούλιο, η υπογραφή και η αποστολή στο Κοινοβούλιο να γίνει κάποια στιγμή το 2015. Ο ρυθμός ήταν ιδιαίτερα ταχύς και δύσκολος. Η Επιτροπή λοιπόν ε, είναι περήφανη για το έργο της και προσβλέπει στην στήριξη και των συνομοθετών, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερη απασχόληση και θέσει εργασία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Πρώτο ομιλητή, η πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Κρίστα Ρόβολ, δεν έχει ε, ακόμη φτάσει. Οπότε θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Σαλβατόρε Τσίκα, πρώτο ομιλητή του ΕΛ, για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως οι πτυχές που ανέφερε ο Επίτροπος είναι σημαντικές όσον αφορά όλος ιδιαίτερος τις προσδοκίες που είχαμε ε, για αυτή την συμφωνία. Μια συμφωνία που την έχουμε μελετήσει, την έχουμε ε, δουλέψει και που βέβαια ε, προκαλούσε το θέμα της διαφάνειας και της προστασίας της μικρομεσαίας μας επιχείρησης αλλά και το άνοιγμα μιας μεγάλης αγοράς. Πιστεύω πως έγινε το έργο και πιστεύω πως έγινε το έργο διότι πάνω απ' όλα στη διαδικασία της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την προστασία των ε, γεωγραφικών ενδείξεων επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα που είναι σημαντικό και που ε, αναγνωρίζει 125 από τις 145 γεωγραφικές ενδείξεις ε, να προστατεύονται, να είναι εγγυημένε και να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, σε μια διεθνή αγορά πολύ σημαντική. Θα ήθελα να κάνω, ωστόσο, να αναφέρω μάλλον έναν προγραμματισμό για αυτή την πτυχή. Πιστεύω πως είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να κληθεί να δώσει τα μέσα, να, δώσει, να παίξει έναν καθοδηγητικό ρόλο και να συνοδεύσει τη διαδικασία συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή την ε, ε, προσπάθεια, ακριβώ διότι λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών τους δεν είναι κατάλληλες για να ε, μπορέσουν να υλοποιήσουν με συγκεκριμένο τρόπο άμεσα μάλλον να κατανοήσουν αυτούς τους κανόνες, αυτά τα προγράμματα και αυτές τις συμφωνίες. Για να υπάρξει λοιπόν μια αποτελεσματική ε, παραγωγή και ένας αυτοματισμός, οφείλουμε με κάθε κρατος να δημιουργήσουμε αυτές τις δυνατότητες, να υπάρξει ένας ε, ε, σπόνσορας, ένας χορηγός, ένας καθοδηγητής, γιατί είμαστε σε φάση κρίσης όπου οι μικρομεσαίες κλείνουν, όπου οι περιφέρειες αφήνονται στη μοίρα τους και να προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα μπορέσουν να βγουν από τα προβλήματα. Πιστεύω πως είναι σημαντική λοιπόν η συμφωνία αυτή που επετέθη, αλλά δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο με ευαισθησία και με οραματισμό να δώσουμε συγκεκριμένες διαστάσεις σε αυτό το ρόλο του ανοίγματο της αγοράς σε μια Ευρώπη που χρειάζεται στις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξαναβρει την αξιοπρέπεια, τη δυνατότητα, μια διέξοδο που σίγουρα μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί εξάλλου θα ήθελα να προσθέσω και πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι ο κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων δεν είναι οριστικός, δεν έχει κλείσει. Υπάρχει ακόμα δυνατότητα, πέρα του να έχουμε το παρμεζάνα, να έχουμε για παράδειγμα που εγώ προέρχομαι από τη Σαρδινία, το πεκορίνο της Σαρδινίας ή της ε, Ρώμης, περιοχής της Ρώμης. Θα έπρεπε δηλαδή να μπουν και άλλες ε, γεωγραφικές ενδείξεις και άλλες προστασίες εγγύησης, δυνατότητες και ευκαιρίες για τις ε, περιφέρειες που χρειάζονται αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με αυτό το σύστημα το οποίο υποφέρει να βρουν μια άλλη διέξοδο. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίκου. David Μάρτιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ. Για τη συμφωνία αυτή έχω ερωτήσεις και σχόλια. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι σίγουρος ότι το Συμβούλιο θα προχωρήσει στην υπογραφή. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Είναι για πολιτικούς λόγους, είναι γιατί έχει αντιρρήσεις επί του κειμένου ή θεωρεί το Συμβούλιο ότι το κείμενο το ικανοποιεί. Τώρα, αν ολοκληρωθεί οι επενδυτές πώς θα δουν το διαπραγματευμένο αυτό κείμενο. Όπως ξέρετε κύριε Επίτροπε, η ομάδα μου θεωρεί πιο εύκολο να μπει και να συμφωνήσει με τη συμφωνία αυτή αν αφαιρεθούν τα επίμαχα ζητήματα. Για τα φάρμακα, για παράδειγμα, ακούσαμε από τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων να μας, δίνει, να μας κάπως, αλλά θα ήθελα να το ακούσω και από εσά κύριε Επίτροπε, ότι η συμφωνία αυτή δεν θα πλήξει την αγορά των ε, φαρμάκων αυτών που πηγαίνουν στον τρίτο κόσμο. Επίσης, όσον αφορά την απαγόρευση διοξεδίου του άνθρακος ή άλλα θέματα και ακόμα και αν είναι χωριστά από την εμπορική συμφωνία, θα ήθελε ο Επίτροπος να μας πει ότι εξακολουθούν να δουλεύουν για να σωθούν αυτά τα ζητήματα ακόμα και εκτός συμφωνίας. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όπως και ο Επίτροπος, βλέπω πολλά θετικά μέσα στην εμπορική αυτή συμφωνία με τον Καναδά. Τη γεωγραφική ένδειξη, για παράδειγμα, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πρόσβαση στα γαλακτοκομικά, η... τα ενοπνευματόδη. Καλά, ναι αυτά. Και το ξέρουμε στην ομάδα μου. Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις εννοείται ότι πρέπει να καταλήξουν σε υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Αλλά είναι και μερικά θέματα για τα οποία δεν θέλουμε να κάνουμε υποχωρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν. Επόμενο, επόμενος ο κύριος Τόμασιτς. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Ήδη είπαμε ότι τα τελευταία μέτρα που πήρε η Ρωσία για τα γεωργικά προϊόντα μας δημιουργούν προβλήματα. Και δεν είναι οι τελευταίες τις ενέργειες της Ρωσίας. Αυτό αποδεικνύει τι ζημιά μπορεί να γίνει από την συγκέντρωση των προσπαθειών μας σε κάποιες μεγάλες αγορές. Όμως τα προβλήματά μας με τη Ρωσία δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να προωθήσουμε τις σχέσεις σας με μια άλλη μεγάλη οικονομική δύναμη και ελκυστική αγορά, τον Καναδά. Η συμφωνία αυτή θα ανοίξει για πρώτη φορά την αγορά δημοσίων προμηθειών του Καναδά στους Ευρωπαίους. Θα αυξήσει το εμπόριο και στις υπηρεσίες. Κατά 23% θεωρούμε. Άρα αυτό θα βοηθήσει τη μείωση της ανεργίας και την Ένωση γενικότερα. Γενικότερα αυτό είναι θαυμάσια νέα για την Ευρώπη που χρειάζεται νέους εταίρους. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτή η διαδικασία για την επίλυση των διαφορών δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένους, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί ήδη εννέα κράτη-μέλη έχουν τέτοια διαδικασία επίλυση διαφορών, συμπεριλαμβανομένε και τη Κροατία, στι διμερεί συμφωνίε με τι ΗΠΑ και δεν μα έχουν δημιουργήσει προβλήματα αυτέ οι διαδικασίε διαιτησία που δεν μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα που να μας κάνουν να θεωρούμε ότι θα καταστρέψουν τις οικονομίες μας. Ε, προσπαθεί αυτή η διατησία να ε, ισορροπήσει τα δικαιώματα του κράτους από τη μία μεριά όπου γίνονται επενδύσεις και τα δικαιώματα των ξένων επενδυτών από την άλλη. Η διαδικασία αυτή, ISDS, δεν δίνει υπερβολικά δικαιώματα στον ξένο επενδυτή έναντι της εθνικής κυριαρχίας όπως φοβούνται ορισμένοι. Απλώς διασφαλίζει το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων φυσικά δεν είναι να εμποδίζουν ε, τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αντίθετα, διασφαλίζοντας ε, θεμητό ανταγωνισμό, αυτή η διαδικασία θα συμβάλλει στην ε, δημιουργία κέρδους για τους ιδιωτικούς επενδυτές διότι οι ιδιωτικοί επενδυτές θα είναι πεπισμένοι ότι και αγορές θα παίζουν σωστά το ρόλο τους. Ευχαριστώ κυρία Τόμασίτσου. Έχει ζητηθεί από τον κύριο Λάιχτφριντ μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Κύριε Λάιχτρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι πολύ καταρχάς που σας βλέπω να προεδρεύετε. Είπατε πως δεν δημιουργεί προβλήματα η διαδικασία διαιτησίας. Γνωρίζετε ότι ακριβώς μια ε, ε, καναδική μεγάλη εταιρεία υπάρχει κίνδυνος να ε, διωχθεί από το Ρωμανικό κράτος γιατί δεν είναι δεδεθμένο το Ρωμανικό κράτος να ε, δεχθεί να εκδιωχθούν κάποιοι πολίτες και σε άλλες περιπτώσεις διάφορα κράτη στρέφονται κατά διεθνών εταιριών. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν δημιουργεί προβλήματα αυτή η διαδικασία διατησίας. Κυρία Τόμασιτς, 30 ε, δευτερόλεπτα. Μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, λέει η κυρία Τόμασιτ, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλων διαστάσεων που να θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία. Χάσαμε τη Ρωσία. Αν πρόκειται να χάσουμε τον Καναδά, τι αγορέ θα βρούμε. Μπορούμε να έχουμε αρχέ, αλλά δεν θα έχουμε θέσει εργασία. Ευχαριστώ. Η Μαρίτε Σάκε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων το να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή με τον Καναδά είναι μεγάλο επίτευγμα. Συγχαρητήρια και για την Ευρώπη και για τον Καναδά. Ελπίζω να είναι μια συμφωνία από την οποία όλοι να έχουμε να κερδίσει. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί κάνουμε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες, γιατί βοηθούν την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Ιδίως μάλιστα τώρα που η Ρωσία έχει αντιδράσει όπως αντιδράει στις κυρώσεις που βάλαμε εμείς. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν που έχουμε για να ελαφρύνουμε λιγάκι τη ζημιά για τις επιχειρήσεις μας είναι να διευκολύνουμε τις εξαγωγές και να βρούμε άλλες αγορές αλλού στον κόσμο. Η πρόσβαση στις ε, προμήθειες είναι κάτι που περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή και βελτιώνονται οι προδιαγραφές για την ε, διατροφική ασφάλεια. Το πιο επίμαχο βέβαια είναι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 1.400 τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες διαμάχες όπου δεν διέπει το κράτος δικαίου. Ενώ τώρα αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχει μεγαλύτερη αμεροληψία από τους διαιτητές και καλύτερη προστασία σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά το βασικό κλειδί είναι το κατά πόσο χρειαζόμαστε το ISDC μεταξύ δύο δημοκρατικών χωρών. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Και είναι κάτι που τίθεται όχι μόνο για την εμπορική αυτή συμφωνία με τον Καναδά, αλλά και για άλλες περιπτώσεις, γιατί μήπως πρέπει να βρούμε κάποια άλλη λύση για τέτοιες εταιρικέ σχέσεις που διαπραγματευόμαστε υπερατλαντικά. Πολύ θα ήθελα να ξέρω περισσότερα επίσης για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, όπου συμμετείχαν πολλοί πολίτες. Παρόλο λοιπόν που το κείμενο της συμφωνίας αυτής δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προβεί σε αναθεώρηση πριν καταλήξουμε οραστικά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρή Μινέρ για μισή λεπτό. Ah, dat werkt, dank u. Voorzitter, het Πρόεδρε, η συμφωνία ΣΕΤΑ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και αυτό το θεωρούμε καλή είδηση. Είναι πολλά ακόμη τα εκκρεμή ζητήματα στα οποία θα, τα οποία θα πρέπει να κρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δίνει υπερβολικά πολύ ισχύ εξουσίες στις μεγάλες επιχειρήσεις και στην καναδική πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από πλευράς ε, των πολιτών που όμως αγνοήθηκαν. Πολιτών που ψήφισαν για το κοινοβούλιο. Πολιτών που κύριε Ντεχιούχτ είναι τα αφεντικά σας. Είναι προφανές ότι οι πολίτες της Ένωσης δεν θέλουν μια τέτοια συμφωνία, δεν θέλουν μια τέτοια συνθήκη, δεν θέλουμε να υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, μπορούν να ανατρέψουν την υφιστάμενη δημοκρατία και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Δεν ε, βλέπω λοιπόν αν μπορείτε να μας δώσετε εγγυήσει ότι δεν θα παραβιαστεί η δημοκρατία. Έχετε τέτοια δυνατότητα να εγγυηθείτε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα είναι σε θέση να λάβουν απόφαση για εγκατάλειψη της πυρηνικής επιλογής χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από διαιτησία ή από διαδικασία επίλυσης ε, διαφορών στο πλαίσιο της ΣΕΤΑ. 16 ευρωπαϊκά κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου και του Ολλανδικού, σας απέστειλαν επιστολή όπου λένε πως οι συμφωνίες όπως η TTIP και η ΣΕΤΑ πρέπει να παραμείνουν μικτού χαρακτήρα συνθήκες προκειμένου να έχουν λόγο και τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό. Παρακαλώ να τελειώνετε, λέει ο Πρόεδρος. Η ΣΕΤΑ και η ΤΙΤΙ πρέπει να παραμένουν μεικτού τύπου συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ζαντού για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Προφανώς για τους οικολόγους η συμφωνία αυτή για την οποία θα ενημερωθούν οι πολίτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει, χωρίς όμως να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων αυτών. Αυτή η συμφωνία έχει, ενέχει πολύ περισσότερους κινδύνους από ό,τι ωφέλει, ιδιαίτερα για τη γεωργία όπου έχουμε να κάνουμε με εκμεταλλεύσεις καναδικές δεκαπλάσιου μεγέθους κατά μέσο όρο από αυτές της Γαλλίας, με κινδύνους γνωστούς σε σχέση με την κτηνοτροφία. Για το θέμα των ε, γενετικά τροπημένων οργανισμών φαίνεται να προκύπτει μέσα από τη συμφωνία ένα φόρουμ συνεργασίας μεταξύ καναδικών και ευρωπαϊκών αρχών συμπεριλαμβανομένου και του στόχου της ε, μη ανατροπής από τις ευρωπαϊκές αρχές των προοπτικών για ε, εμπορικές συναλλαγές. Εμείς θεωρούμε ότι η τη Συμφωνία δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο ως εμπορικό εργαλείο, αλλά ως εργαλείο υποστήριξης κυρίως των τοπικών ε, επιχειρήσεων και ιδιαίτερα το ζήτημα του ESDS, βλέπετε ότι η ΣΕΤΑ, ε, βλέπετε ότι όλο και τον κόσμος, πολίτες αλλά και εδώ το Κοινοβούλιο αμφισβητεί αυτή τη συνθήκη διότι η ίδια η συνθήκη έχει ανατρέψει τη δυνατότητα της λήψης αποφάσεων από τον πολίτη και το Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ανατρέψει τη συμφωνία αυτή κυρίως όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρεών ή τραπεζών. Για μας όμως αυτό δεν θα αρκέσει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αρκέσει και γι' αυτό ε, ελπίζω όλοι όσοι σήμερα τοποθετούνται κατά τη συμφωνία αυτή να διατηρήσουν την αντίστασή του τι επόμενε ημέρε. Πρέπει η ΣΕΤΑ να απορριφθεί και ιδιαίτερα όσον αφορά τι επενδύσει. κυρία Τετιάνα για λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως και η TTIP είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει με μυστικότητα στις αίθουσες των Βρυξελών και αποφασίστηκε από γραφειοκράτες που δεν τους έχει εκλέξει κανείς και κανείς δεν είναι υπόλογος για αυτό που κάνει. Ακριβώς όπως και για την TTIP ε, θα είναι άγνωστες οι συνέπειες και στη συμφωνία με τον Καναδά. Διότι η μείωση των, ε, και άρση των δασμών δεν αρκεί. Ε, αυτό γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν αρκεί για να απολυθεί ένα προϊόν σε μια χώρα που έχει τελείω διαφορετικές, ε, ε, διαφορετικούς κανονισμούς. Ξέρετε λοιπόν τι σημαίνει να έχουμε γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς ε, στο τραπέζι μας και φυσικά ο Καναδάς δεν τηρεί και τους όρους που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Καναδάς δεν έχει προσπογράψει και την παράταση του πρωτοκόλλου του Κιώτου. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και ξέρω τι σημαίνει να παράγει κάποιος ένα προϊόν με περιβαλλοντικά πρότυπα και άλλα πρότυπα όπως πρέπει για μα εμά, με τα οποία είμαι σύμφωνη. Τι θα γίνει όμω με όλου αυτού οι οποίοι δεν υποχρεωμένοι να σεβαστούν όλα αυτά τα θέματα. Και αναφερόμαστε στο περιβάλλον όταν στον Καναδά, στην περιοχή τη Αλβέρτα, ε, γίνεται εξόριξη πετρελαίου από. Ε, Αγωγού, ε, αποψηλώνοντα ολόκληρα δάση. Πραγματικά με αυτή τη συμφωνία θα υπάρχει μεν πρόσβαση σε φθηνότερο πετρέλαιο, αλλά το τίμημα ποιο θα είναι. Και επίση, το ISDS πρόκειται για μια ρήτρα η οποία πραγματικά θα ήταν γελία εάν δεν ήταν τόσο επικίνδυνη. Επιτρέπει σε μια πολυεθνική να προσφύγει κατά κάποιου κράτους. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, απευθύνομαι σε εσά. Με μια δημόσια ακρόαση η οποία έγινε όταν όλα ούτω ή άλλω διακόπτει ο πρόεδρο στην ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Λεπέν. Θα συνδώσω, θα εκτείνω την προηγούμενη ε, παρέμβαση. Η συμφωνία αυτή θα ψηφιστεί σύντομα εδώ. Ένα κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, αυτό της δικαιοσύνης. Το κείμενο προβλέπει μια ιδιωτική δικαιοσύνη μεταξύ ε, κρατών και πολυεθνικών εταιριών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ε, διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών ε, πρόκειται για μια ε, διατητική ε, διαδικασία που θα κινητοποιείται όταν μια πολυεθνική εγκαταστημένη στη Γαλλία δεν, τη δεν της αρέσουν οι νόμοι της Γαλλίας. Θα είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπέρ των συμφερόντων των πολυεθνικών μια τέτοια ε, περίπτωση μπορεί να είναι ε, να έχει σχέση με, μια, ε, σχιστο, με, με επενδύσεις, κανονικές επενδύσεις, σχιστολιθικό αέριο, ε, οι οποίες θα κρίνονται κατά βάση από ιδιωτικά δικαστήρια. Η, δια, η δικαιοσύνη όμως θα πρέπει να είναι δικαίη και διαφανής. Είναι η μοναδική εγγύηση που μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες μας σχεδόν ε, όλοι οι ε, βουλευτές ε, στο διεθνές επιμελητήριο, εμπορικό επιμελητήριο των Βρυξελών κατέθεσαν την αντίθεσή τους. τώρα θα πρέπει να ψηφίσουν και να ψηφίσουν αρνητικά γιατί είναι πραγματικά ντροπιαστικό αυτό που μας προτείνει η Κομισιόν. Γιατί δεν πρόκειται για δικαιοσύνη, πρόκειται για αδικία. Τουλάχιστον δείξτε γενναιότητα μία φορά. Ψηφίστε όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπέν. Τρία λεπτά. Ο κύριος Προύστ. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ε, κυρία Λεπέν, νο, σας ακούει κανείς και νομίζω ότι είναι τραγική κατάσταση. Σαν να ε, νομίζετε ότι ε, ε, χωρούμε τα πάντα στην ε, Κομισιόν. Δεν είναι έτσι. Ασφαλώς πρέπει να κρίνουμε και να επικρίνουμε αλλά με επιχειρήματα. Ε, αυτή τη στιγμή ανακατεύεται επιχειρήματα με συνομωτησιακές θεωρίες. Ε, προσπαθείτε να κρίνετε πολύ υπερβολικά νωρίς. Κάποιοι κλούν τον κόντρα του κινδύνου αδίκως. Ασφαλώς και πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία με μια δυτική χώρα, σύμμαχο χώρα. Ασφαλώς και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, γιατί δίνουμε μια εντολή στην Κομισιόν και πρέπει να τη φέρει σε πέρας, σε πέρας. Δεν θα πρέπει να ξεπεράσει την κόκκινη για τις κόκκινες ζάμες μας. Όμως πάνω απ' όλα θα πρέπει να εξηγήσουμε τόσο σε ό,τι αφορά τον Καναδά όσο και αργότερα τις ΗΠΑ ε, και δεν θα πρέπει να ε, διεκτραγωδούμε την κατάσταση. Συμφωνούμε, ε, υπογράφουμε μια συμφωνία ελεύθερων ε, ανταλλαγών ε, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε την επιθετική πολιτική της Ρωσίας, εμπορική πολιτική της Ρωσίας. προσπαθούν να, ε, προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ε, είμαστε δολοφόνοι της, ε, ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας ή δεν είμαστε δημοκράτες. Όμως για αυτά χρειαζόμαστε, χρειάζεται πιο συγκεκριμένα επιχειρήματα. Ο, οι άνθρωποι χρειάζεται να καταλάβουν ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποφέλθουν από αυτές τις συμφωνίες, να ανοίξουν καινούριες αγορές. Οι επιχειρήσεις μας θα έχουν ισότιμη ε, πρόσβαση στην αγορά του Καναδά. Κάποιοι όμως περιμένουν ένα όχι του Κοινοβουλίου ε, για να κλείσουν το δρόμο προς μια οποιασδήποτε πρόοδο σε αυτήν την κατεύθυνση. Πώς θα μας εγγυηθείτε κύριε Επίτροπε ότι θα τύχουν σεβασμού αυτές οι συμφωνίες. Με ποιο, ποια είναι τα μέσα ε, που διαθέτεται για να παρακολουθείτε την υλοποίησή τους. Και ποιες είναι οι εγγυήσει τελικά έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο Καναδάς θα εφαρμόσει αμοιβαία αυτή τη συμφωνία και δεν θα ε, δίνει προνόμια στις δικές του επιχειρήσει εναντί των δικών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προύστ και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Λάνε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με τρία θέματα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία με τον Καναδά. Καταρχάς, κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι έχουν γίνει πολύ επικριτικές συζητήσεις σε πολλούς κύκλους της κοινωνίας των πολιτών στην, Ευρά, στην Ευρώπη και πρέπει να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο στις 6 Αυγούστου να λαμβάνει μόνο το κείμενο και γιατί δεν έχετε δημοσιεύσει ακόμη το κείμενο. Μας λέτε ότι σε μερικές μέρες θα το δημοσιεύσετε. Εγώ νομίζω ότι για να υπάρξει λογική συζήτηση και σε επίπεδο κοινή γνώμη πρέπει εγκαίρως και πολύ σύντομα να δημοσιευθούν τα κείμενα για να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να τα μελετήσουν και να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι, βεβαίω θα υπάρξουν κάποια πολύ θετικά στοιχεία τα οποία διαβλέπω εγώ με βάση παραδείγματι το θέμα των γεωγραφικών δικτών για την γεωργία, για την πρόσβαση στην αγορά, καμία αμφιβολία προς αυτό, αλλά ε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο οι ρήτρε standstill και άλλες θα επηρεάσουν την παροχή των υπηρεσιών στην περίπτωση αυτή. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε πολύ προσεκτικά. Και το τρίτο σημείο, κύριε Επίτροπε, έχει να κάνει με τον μηχανισμό ε, προστασίας των επενδύσεων, επίλυση διαφορών. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα πρόσβαση σε ένα τέτοιο μέσο. Είχε αυτό σχεδιαστεί σε ένα μηχανισμό διαφύλαξη διασφάλιση έναντι κρατών που θα είχαν ενδεχομένω μη δημοκρατικέ δομέ. Εδώ βλέπουμε να στρέφεται κατά δημοκρατικών αποφάσεων κοινοβουλίων. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εποχή στην οποία ζούμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοιο μηχανισμό. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις και να μεριμνήσετε έτσι ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα ε, ικανοποιητικό για να μην έχουμε ένα δεύτερο άκτα. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Ένα λεπτό ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ένα από τα συνεχιζόμενα ε, στοιχεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συμφωνία TTIP η οποία φυσικά επικεντρώνει και την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, και φυσικά η συμφωνία με τον Καναδά ε, δεν υπολείπεται. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίω στο γεωργικό τομέα, γιατί οι συνάδελφοι μίλησαν για διάφορου άλλου τομεί. Ο γεωργικός τομέας είναι ο τομέας ο οποίο θα πληγεί περισσότερο. Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή είναι μία από τις πιο φιλόδοξες ε, συμφωνίες στο γεωργικό τομέα. Οι παραγωγοί ε, τοπικά θα έχουν κάποιες ελπίδες ε, από τις αναγνωριμένες γεωγραφικέ ενδείξει και τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και θα υπάρχει και προστασία της ε, μεγάλης πλειονότητας αυτών των γεωργών. Αυτό είναι πτυχές της συμφωνίες, στις ε, οποίες θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσει και θεωρώ ότι σηματοδοτούν και το μέλλον των εμπορικών συμφωνιών. Ε, κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τοπικούς γεωργούς και παραγωγούς και σας ε, ε, λέω ότι ανησυχούν εξίσου με αυτή τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και εμείς ανησυχούμε και θεωρώ ότι σε όλες τις συμφωνίες υπάρχει ένας βαθμός υπερβολής στα όσα μπορεί να, συμβούν ή να μην συμβούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε εμπιστοσύνη και να αντλήσουμε διδάγματα από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίκολσον. Για ένα λεπτό κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Ντεγκούχιτ. 500.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουν αντιδράσει στο θέμα των διαβουλεύσεων του ε, μηχανισμού επίλυσης που έχετε παρουσιάσει ως κομμάτι της συμφωνίας ΣΕΤΑ. Πριν όμως μας παρουσιάσετε τη συμφωνία, ε, ε, ακόμα μας λέτε ότι έχουν κλείσει οι διαπραγματεύσεις, ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Και άρα φαίνεται ότι προσπαθείτε να προστατεύσετε τις ε, κερδοσκοπικές αγορές χωρίς κανένα σχεδιασμό για επενδύσεις, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και πάνω απ' όλα καμία δυνατότητα προστασίας ή περιορισμού της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Ε, ούτε των συμβάλλοντων μερών. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες καταστρέφουν την ευρωπαϊκή πολιτική και πρέπει πλέον να αναλάβουμε άλλον δρόμο. Οι πολίτες δεν θέλουν ESDS, ούτε ΣΕΤΑ, ούτε TTIP και εμείς ως δημοκρατικά εκλεγμένοι πρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε τη ΣΕΤΑ ούτε την TTIP. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτς. Ο κύριος Ράιμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν είστε υποχρεωμένο να δημοσιεύσετε την επόμενη εβδομάδα την ε, συμφωνία αυτή, γιατί θα δημοσιεύσει η κοινωνία των πολιτών και φαντάζομαι τι είδου ε, αντιδράσει θα προκύψουν με αυτό το γεγονό Πρόκειται για ένα πολιτικό σκάνδαλο και σκάνδαλο της ε, πολιτικής το γεγονό ότι χρειάζεται η κοινωνία των πολιτών να δημοσιεύσει τη συμφωνία αυτή. Τώρα μα ε, καλείται να λάβουμε απόφαση για να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή, η οποία σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορούμε να λαμβάνουμε καμία απόφαση και να αντιδρούμε σε θέματα που θα έχουν ακόμη και με την υποβολή προσφυγών ει βάρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε να κάνουμε παραβίαση του Ευρωπαϊκού των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δυνατότητα λήψεω αποφάσεων δημοκρατικά από αυτό. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο, να απορριφθεί αυτή η συμφωνία και δεν βλέπω καμία άλλη δυνατότητα ε, δράσεως για μας, τους εκπροσώπους, τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η επιλογή σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων ή συγκάλυψης των στοιχείων. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Ράιμον. Ο κύριος Βούλφ έχει τον λόγο. Πρόεδρε, εμείς στο UKIP πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο. Ε, θέλουμε να σχετιζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, δεν είμαστε απομονωτικοί ούτε προστατευτικοί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση είναι ένα, μια προστατευτική τρονιακή ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενιαία αγορά ε, με πολύ ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο. Ε, εμείς υποστηρίζουμε τις αρχές και τις ιδέες πίσω από μια τέτοιου συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ε, που έρει τους εμπορικούς και δολιακούς φραγμούς. Επί της αρχής λοιπόν είμαστε υπέρ. Αναγνωρίζουμε όμως ότι όσο συζητείτε και ελέγχεται πίσω από την αυλαία από ιδιωτικούς φορείς αυτή η συμφωνία θα δημιουργεί προβλήματα. Το δικό μας εκλογικό κοινό ε, φοβάται ότι ε, μπορούμε να διατρέξουμε κίνδυνο από ε, εταιρείες που μπορεί να προσφύγουν κατά τις κυβέρνηση αν θελήσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας. Αυτό δεν είναι σωστό, ούτε δίκαιο. Πιστεύουμε ότι πρέπει κάθε ε, κράτος, έθνος κράτος να μπορεί να φροντίζει το δικό του λαό. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε τέτοιες συμφωνίες. Ε, δεν ε, πιστεύουμε στην ελευθερία, τη δημοκρατία και στο κράτος, έθνος κράτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ούλφη. Κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή την ε, συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρώπης και θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για τα όσα έχει κάνει και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κύριο Μπράτμπουρν, ο οποίος ήταν ε, πρόεδρος της Ορμόδιας Επιτροπής. Θεωρώ ότι ήταν ε, πολύ καρποφόρο το αποτέλεσμα και αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει στο μέλλον. οποιαδήποτε συμφωνία με τον Καναδά είναι απόλυτα λογική, γιατί ο Καναδάς είναι ιστορικά πιο κοντά σε εμά από πλευράς πολιτισμού, γλώσσας, ε, Νομοθεσία και πολιτική. και μπορεί να διήρκησαν πέντε χρόνια οι διαπραγματεύσει για αυτή τη συμφωνία. Θεωρώ όμω ότι καταλήξαμε σε μια λογική συμφωνία εν τέλει. Υπάρχουν βεβαίω δυσκολίε οι οποίε επισημάνθηκαν ε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να την υποστηρίξουμε ε, ταυτόχρονα εκφράζοντα και τι επιφυλάξει μα. Γι' αυτό το σκοπό απέστειλα μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκφράσω την ανησυχία μου για την ε, ε ε, η εισαγωγή του βόηου κρέατος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω το, ο τομέας του βόηου κρέατος να αναγνωριστεί ως συγκεκριμένο τομέας, γιατί ο τομέας του βόηου κρέατος είναι μικρής ε, κλίμακας ποιοτικής παραγωγής που βασίζεται στο οικογενειακό μοντέλο γεωργίας και κτηνοτροφίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περιοχή μου αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει τη διάκριση μεταξύ υψηλής ποιότητας ε, κρέατα, ε, κρεάτων κοπής ε, συγκεκριμένης και ε, χαμηλότερης ποιότητας και ότι τα υψηλής ποιότητας θα μπορέσουν να είναι εξαγωγές οι οποίες θα είναι πολύ ποιοτικέ και θα είναι πολύ λογικές όταν θα φτάσει και η εποχή του μπάρμπεκιου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ε, Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να εκφράσω και την ε, ε, δυσαρέσκειά μου ε, για τη ρήτρα αναθεώρησης διότι αν όπως αναμένω υπάρξουν δυσκολίες ε, από αυτή την ε, ρήτρα αναθεώρησης ε, θα δημιουργηθούν προβλήματα και φυσικά αυτή η ρήτρα πρέπει να λεφθεί υπόψη και για την TTIP γιατί η TTIP δεν θα μπορούσε να λάβει υπόψη της αυτό το στοιχείο που έχουμε για το βόλιο κρέας θα αλλάξουν τα πράγματα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επταπλάσια προβλήματα. Οι λεπτομέρειες λοιπόν αυτά έφτασαν ε, στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο στις 25 Αυγούστου. Μπορεί εγώ να μην είμαι τόσο να είμαι προνομιούχος, δεν ξέρω αν οι άλλοι έλαβαν γνώση. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Δύο λεπτά ο κύριος Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε πίτροπε. Στις ε, εθνικές εκλογές στην Αυστρία εμφανίστηκε μια λίστα εκλογική από έναν εκατομμυριούχο, ο οποίος στα δισεκατομμυριά του τα έκανε σε μεγάλο βαθμό στον Καναδά και ο οποίος σε σχέση με την... Ε, όταν το ρωτήσανε σε σχέση με τις ε, ε, απόψεις του για τη δημοκρατία είπε ότι ισχύει ο χρυσούς κανόν. Όποιος έχει στα χέρια του το χρυσάφι κάνει και τους κανόνες. Τον ακούσαμε λοιπόν, γελάσαμε, δεν τον πήραμε και πολύ σοβαρά. Τώρα όμως, όταν κοιτάω αυτά τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με τη συμφωνία με τον Καναδά αλλά και με τι ΗΠΑ δεν είμαι βέβαιο αν θα πρέπει να κλαίω, να γελάω ή αν θα πρέπει σιγά σιγά να φοβάμαι ότι τελικά αυτό πραγματι... πραγματοποιείται. Και προσπαθώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να περιμένετε ότι η δημοκρατία η ευρωπαϊκή δεν θα έχει σοβαρέ επιφυλάξει για μια τέτοια συμφωνία. Δεν θα τη βλέπει δηλαδή ω ένα σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατία και για το κράτος δικαίου. Το να μπορούν να ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπαγωγής στα εθνικά δικαστήρια ή στην δικαιοδοσία την κρατική οι μεγάλες επιχειρήσεις όταν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες ε, αποφασίζονται από τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε έξω από τις δημοκρατικές διαδικασίες πράγματα τα οποία πειράζουν τους τη ζωή τους. Εδώ υπάρχουν και πρωτοβουλίες πολιτών τις οποίες αγνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι μη δημοκρατικό. Έχουμε να κάνουμε πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα και όπου έχουμε φτάσει στο σημείο να εκφράζεται μία πλειονοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία ενδέχεται να καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία παρά τα θετικά της στοιχεία. Θέλετε λοιπόν να καταρριφθεί αυτή η συμφωνία, να απορριφθεί. Εκεί θέλετε να καταλήξει αυτή η συμφωνία. Δεν θα έπρεπε να προσπαθήσετε να επιτύχετε τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για να συζητηθεί αυτή η συμφωνία. Γιατί αν δεν υπάρξουν δεν θα συζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάιφτριτ. Η κυρία Φορέντσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και σήμερα η συζήτηση για την Συμφωνία ΣΕΤΑ αναφέρθηκε σε οικονομικά ωφέλη και την ανάγκη αυτής της συμφωνίας. Ε, στην ε, πραγματικότητα, σε αντίθεση με την ε, TTIP, της οποίας είναι ο πρόδρομος, ε, προσπαθεί να θέσει τα ιδιωτικά συμφέροντα υπέρ της ε, οικονομικής βιωσιμότητας. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε ενώπιον μια συμφωνίας ε, χωρίς καμία παρακολούθηση από την κοινή γνώμη και όπου τα πάντα γίνονται με πάσα μυστικότητα. Οι κοινωνικές πτυχές της συμφωνίας θα πρέπει να μας ανησυχούν και το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ε, εγγύηση για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αγορά εργασίας. Για άλλη μια φορά πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ουσιαστικά δρούν για να αποδυναμώσουν το σύστημα της εργασίας και στην Ευρώπη και στον Καναδά εις βάρος ε, των ε, εργαζομένων και υπέρ του κέρδους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπάθησε να τηρήσει τα πρότυπα εργασίας και πρόνοιας και εμείς δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση και εντός και εκτός αυτού του κοινοβουλίου θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία κατά τη συμφωνία ΣΕΤΑ όπως και όλες τις συμφωνίες όπως η TTIP διακόπτει ο Πρόεδρος Νομιλίτυπα. Ευχαριστώ κύριε Φορέντσα για ένα λεπτό ο Σάνφος κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως ε, πράσινος ευρωβουλευτής ε, ε, καλό να απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή. Κυρίως διότι ε, περιέχει ένα βλαβερό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που πλήττει και τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Η διαβούλευση την οποία διοργάνωσε η Κομισιόν για μια, ένα παρόμοιο σύστημα στη συμφωνία TTIP ε, έδωσε 150.000 απαντήσεις τις οποίες ακόμα αναλύει η Κομισιόν φαντάζομαι. Γιατί λοιπόν ε, η συμπερίληψη αυτής της, αυτού του συστήματος εδώ, σε αυτή τη συμφωνία ε, έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτές οι αντιδράσεις. Αν ο μηχανισμός ISDS παραμείνει στην ΣΟΕΣ ε, θα πλησιάσουμε κοντά σε, ένα, σε μια κατάσταση όπου οι εταιρείε θα γράφουν το δίκαιο και την νομοθεσία. Οπότε ζητώ από τον David Cameron και τους άλλους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων ε, να απορρίψουν αυτή τη συμφωνία. Αυτό θα κάνουν οι πράσινοι όταν έρθει η συμφωνία αυτή προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Ο κύριος Κόβατσεφ, δύο λεπτά уважаеми господин Κύριε Επιτροπέ, Πρόεδρε, συνάλφοι, πρέπει να διευρύνουμε την συνεργασία μας με τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι στενός, καλός εμπορικός μας εταίρος. Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε βάθυνση των σχέσεων μας. Θα αλλάξει το διατλαντικό χώρο, θα τον καταστήσει μια εμπορική ζώνη. Οι ανταλλαγές θα αυξηθούν κατά 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι οικονομικές μας σχέσεις θα γίνουν πιο στενές και αυτό θα μας οδηγήσει σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Όμως, να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο, στην πρόσβαση στην καναδική αγορά. Αυτή η πρόσβαση θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα σήμαινε την άρση των περιορισμών ε, σε ό,τι αφορά την ε, έκδοση θεωρήσεων για πολίτες ε, χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Ε, δεδομένου το τι συμβαίνει στα ανατολικά μας σύνορα, αυτή η συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί πολύ θετική για την οικονομία μας. Θα πρέπει να εντείνουμε την βορειοατλαντική μας συνεργασία. Επίσης, η ε, επικοινωνιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την Καναδά και τις ΗΠΑ θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να καθησυχαστούν οι ανησυχίες που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε ε, να μην διαδίδονται φημολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόβατσοφ. Η κυρία Αρένα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ οι συνάδελφοι τη ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ήδη υπενθύμησαν μια σειρά από επιφυλάξει που αφορούν τη συμφωνία ΣΕΤΑ και ιδιαίτερα το μηχανισμό απειλή διαφόρων. Δεν θα επανέλθω στο θέμα αυτό λοιπόν. Εγώ κυρίω ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο μηχανισμό ρυθμιστική συνεργασία όπω αυτό προβλέπεται τώρα στην συμφωνία ΣΕΤΑ. Γιατί πρόκειται για ένα μηχανισμό που επιτρέπει σε πολυεθνικέ, όντω και ευρωπαϊκέ αλλά και ε, καναδικέ, να προσδορίζουν μια σειρά από κανόνε που τι εξυπηρετούν και που ως εκ τούτου δίνουν ζωή στην συμφωνία. Δηλαδή η αρχική ε, δέσμευση που ήταν να μην αναθεωρηθούν προς τα κάτω οι προδιαγραφές και οι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα τηρηθούν διότι οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις μεταξύ τους θα μπορούν να αποφασίσουν ότι οι κανόνες ε, που ισχύουν στα κράτη μας αντιβαίνουν στην ελεύθερε στις ελεύθερες Εσείς κύριε Ντεκιούχης είχατε, είχατε πει κάποια στιγμή ότι ασφαλής αξία για σας ήταν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ρυθμίσεις και ότι δεν πρόκειται να υποβιβαστούν, αλλά τώρα βλέπουμε ένα μηχανισμό ο οποίος αμφισβητεί και ανατρέπει τη δέσμευσή σας. Θα ήθελα μια σαφή δέσμευση λοιπόν και τοποθέτηση από πλευρά σας. Υπάρχει όντως η δυνατότητα να διαφυλαχθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ρυθμίσεις σε θέματα ε, δημόσιας υγείας, κοινωνική κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας ή περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρενά. Η ευχαριστω Σάντσες Καλντεντέη. Ένα λεπτό. καλτεντει ενα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, δεν ξέρω αν μας διαφεύγει η επονίδιστη επίθεση ε, στη δημοκρατία, η οποία προκύπτει με αυτή τη συμφωνία και στην οποία συζητάτε όλοι. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει. Το χειρότερο παράδειγμα είναι να δεχτούμε την, ε, ε, θα πρέπει να δεχτούμε την πρωτοβουλία των πολιτών για να σταματήσουν όλες αυτές οι συμφωνίες οι οποίες είναι εις βάρος της λαϊκής θέλησης ξεπουλούν τους Ευρωπαίους. Η συμφωνία αυτή είναι εις βάρος των πολιτών και προς όφελος των επενδυτών και το χειρότερο είναι ότι το γνωρίζουν. Κύριε Επίτροπε, δεν είστε πολιτικοί, είστε άνθρωποι του εμπορίου και έμποροι και δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Θα πρέπει να ε, μιλήσετε ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης για την ε, φορολογική απάτη για την οποία ε, έχουν προσφύγει εναντίον σας. Εμείς προσπαθούμε να προσπίσουμε τα ε, συμφέροντα της πλειοψηφίας των ανθρώπων και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τέλους. Ε, δεν φτάνει που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τη Συμφωνία Άκτα, το ίδιο θα κάνουμε και με τη ΣΕΤΑ. Και θα το δείτε στις 20 Οκτωβρίου σε όλη την Ευρώπη. Διακόπτει την ομιλήτρια ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κυρία Σάντρες Καλεντρή. Η κυρία Κέρτιν Ντόρλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, αλλά σε μια περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον για τις ε, εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες ε, οι ομιλίες περί διαφάνειας και πολιτικής συμμετοχής ε, δεν θα έχουν καμία ουσία εάν δεν τεθούν πραγματικά στην πράξη. Μετά από τα όσα συνέβησαν με το κείμενο της ΣΕΤΑ και τα όσα προχωρούμε με την TTIP η οποία χρησιμοποίησε το κείμενο της ΣΕΤΑ ως ε, ε, πρότυπο, τι μήνυμα αποστέλουμε στους πολίτες. Οι συμφωνίες για τις υπηρεσίες αυτές ε, και οι υπηρεσίες κοινή ωφελία δεν συζητώνται, δεν έγινε καμία δημόσια συζήτηση για τα όσα έχουν συμπεριλάβει οι κυβερνήσει μα στου αρνητικού καταλόγου και δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών κοινή ωφελία και μέσω του και μέσω ε, συγκεκριμένων ε, ε, κανόνων. Θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς απαιτείται από κάθε κράτος μέλος, γι' αυτό ακριβώς ζητούμε να δημοσιεύσετε ακριβώ τι αναφέρει συγκεκριμένη συμφωνία και τι προϋποθέτει για κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κρίστον Δύο λεπτά. Η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τις θετικέ πτυχές με τη συμφωνία με τον Καναδά, η οποία κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελεί και ευκαιρία για το παραγωγικό μας σύστημα διότι έχουμε ένα οικονομικό σύστημα αλλά και κοινωνικό σύστημα το οποίο δεν απέχει και πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό σύστημα. Και υπό το φως της ε, ε, γεωπολιτικής κατάστασης που υπενθυμίστηκε σήμερα και χθε ε, εδώ στην Ολομέλεια θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιήσει ως ενίσχυση της ε, εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους καλύτερους ε, παίκτες παγκοσμίου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει καλό συμβιβασμό σε θέματα γεωγραφικών ενδείξεων και ε, να λαμβάνεται υπόψη και η παραδοσιακή ε, αποξένωση του Καναδά με αυτό το σύστημα. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρίνει με τον καλύτερο δυνατό ε, τρόπο, με πάσα ειλικρίνεια τη συμφωνία αυτή, ε, προσπαθώντας να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στα όσα προβλέπει η συμφωνία και να μην έχουμε ε, μία ε, κατανοητή μεν αλλά επικίνδυνη αλληλοεπικάλυψη με τη συμφωνία TTIP διότι θα χάσουμε τις καλές πτυχές αυτής της διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι πολλά στοιχεία αυτής της συμφωνίας μπορούν να βελτιωθούν ακόμα, γι' αυτό ακριβώς ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν όλες οι δυνατές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μόσκα και τώρα για ένα λεπτό κύριο Σούστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επιτροπέ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε το κείμενο της ΕΤΑ πλέον ε, και πρέπει ε, και από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή θα κηρύξει ότι έχουν λήξει οι διαπραγματεύσει. Αυτό όμω είναι εσφαλμένο χωρί να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εξετάσει επί τη ουσία το κείμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρέ ανάγκε για βελτίωσή του. Η Συμφωνία για την Προστασία των Επενδύσεων σημαίνει την ίδρυση έξω από τα εθνικά ένομα συστήματα διαιτητικών δικαστηρίων ε, που ανατρέπουν μια βασική αρχή ότι δηλαδή οι πάντες είναι ίσοι ενώπιον του ε, νόμου. Ε, κάποιοι θα είναι πιο ίσοι από ό,τι φαίνεται με τη νέα αυτή συμφωνία. Επίσης αρνητικοί οι κατάλογοι για το ποιοι τομείς δεν υπάγονται σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ λίγοι οι τομείς οι οποίοι θα μπορούν να επανακοινωτικοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ανατροπή της δημοκρατικής αρχής και της δυνατότητας αναθεώρησης δεν ε, ικανοποιεί λοιπόν τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου η ΣΕΤΑ. Γι' αυτό καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την αναδιαπραγματευτεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σούστερ. Ο κύριος Μπάλας. Κύριε Επιτροπέ, βλέπετε τη συζήτηση, βλέπετε πώς εξελίσσεται. Ε, δείξτε λίγη σοφροσύνη ο μηχανισμός ISDS δεν πρόκειται να περάσει. Είναι σαφές αυτό. Έγινε μια διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, ε, με την πρωτοβουλία της Κομισιόν ε, και τα αποτελέσματά της δεν ελήφθησαν υπόψη. Αυτό είναι ήδη βαρύ. Δεύτερον, είστε μέλος μιας ε, Κομισιόν η οποία, της οποίας τελειώνει η θητεία. Ο νέος πρόεδρος, ο κ. Γιούνκερ, ε, είπε ότι διαφωνεί με την συμπερίληψη του μηχανισμού ASDS στη Συμφωνία με τις Πολιτείες, οπότε φανταζόμαστε... Εδώ εμείς είμαστε κλεγμένοι ερετοί ε, εκπρόσωποι του λαού ε, και δεν πρόκειται να επιταχύνουμε την διαδικασία προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία αυτή το σύντομο το δυνατό. Καλύτερα να αφήσετε το θέμα αυτό στην επόμενη Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παλάση. Κύριε... Ο κύριος Σίλβα Περέρα. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά είναι μια θετική εξέλιξη. Ε, το οι οικονομικές δυνατότητες που ανήκονται είναι μεγάλες ε, και ε, το καθήκον μας είναι ο συμβασμός να είναι αποδεκτός. Όμω πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση σε, στο πρόβλημα του μηχανισμού ISDS. Είναι ο μηχανισμό επίλυση διαφορών που ε, απειλεί το μέλλον των συμφωνιών όχι μόνο, του, με, το, το όχι μόνο τον Καναδά αλλά και με τι ΗΠΑ και με τον Καναδά και με την Ιαπωνία. Η, Κομισιόν πρέπει να δώσει απάντηση και αυτή η απάντηση πρέπει να είναι πολιτικά βιώσιμη. Οπότε κύριε Επιτροπέ ποια είναι η στρατηγική τη Κομισιόν για το πολιτικό πρόβλημα το οποίο είναι ο μηχανισμό ISDS. Μπορείτε να μας πείσετε ότι ε, η λίστα δοθεί κατά περίπτωση και ότι η ε, ΣΟΕΣ ε, δεν θα είναι πολιτικό, θα αποτελέσει προηγούμενο. Η Κομισιόν μέσω της σύμφωνα της, διαβούλευσης για την TTIP θα δώσει μια συνολική πολιτική απάντηση. Πρέπει η Κομισιόν να δώσει απάντηση, να δώσει μια λύση σε αυτό το θέμα όσο είναι νωρίς κυρία Σίλβα Αυτοί ήταν οι καταγεγραμμένοι ομιλητέ. Περνάμε στη δικασία Καρστιάη. Ο κύριο Σεράου Σάντο. Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στου ιστορικού δεσμού ανάμεσα στον Καναδά και τη χώρα μου, ιδιαίτερα τις Αζόρες. Γιατί στον ε, Καναδά ζουν πολλοί Αζοριάνοι και τα παιδιά τους. Πρόκειται για μια μεγάλη κοινότητα ε, που μάλιστα αντιπροσωπεύεται στην τοπική αυτοδίκηση περίπου 550.000 Πορτογάλοι ζουν στον Καναδά. Σε ό,τι αφορά το, τη συμφωνία ε, και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό, με ένα επίπεδο προστασίας παρόμοιο με αυτό ε, το οποίο ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι ε, γι' αυτό, χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναγνώριση των ε, ονομάτων, των ονομασιών του Τριού, του Σαουζόρζε και του Ανανά των Αζωρών πρέπει την ίδια, ε, στις ίδιες ζήτητες να καταλήξουμε σε άλλες ε, συμφωνίες. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά έχουμε προβλήματα με άλλα θέματα όπως ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε συμφωνίες και σε άλλα μέτωπα, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της ε, δήλωσης του Galway για την ε, παρατήρηση και, την, ε, και τη γνώση σε ό,τι αφορά τον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι ένα κείμενο το οποίο υιοθετήθηκε το 2013 διακόπτει ο Πρόεδρος στον ομιλητή. Σας ευχαριστώ κύριε Σεραοσάντος Η κυρία Χάρκιν. Θα ήθελα στο ένα λεπτό που έχω να αναφερθώ στη συμπερίληψη του ISDS στην ε, προτινόμενη συμφωνία. Και η ερώτησή μου, κύριε Επίτροπη, είναι εξής. Κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ ανεπτυγμένες και έχουν πολύ καλά κατανοητά ε, νομικά συστήματα, γιατί εισαγάγουν τέτοια συστήματα. Και ξέρετε ότι δεν ασυχώ μόνο εγώ. Πάνω από 150.000 πολίτες απάντησαν στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, γιατί όπως και εγώ ανησυχούν για το γεγονός ότι ε, μια επιτροπή διατησία, η οποία θα λάβει την ε, τελική απόφαση δεν θα υπόκειται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ είπε ότι δεν θα δεχτεί η δικαιοδοσία κρατών μελών να περιορίζεται από συγκεκριμένα καθεστώτα για την επίλυση ε, διαφορών επενδύσεων. Και επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ το 2011 σα προειδοποίησε ότι ένα μηχανισμό επίλυση διαφορών κράτου με κράτο και συγκεκριμένα δικαστικά μέτρα είναι τα καταλληλότερα μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, διαφορέ μεταξύ επενδύσεων επενδύσεις. Κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να χάσετε τη συμφωνία. Πριν είναι αργά, θα πρέπει να διαγράψετε τη ρήτρα για το ESDS. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Σέντρα Ρόντριγες τώρα. Ε, Επίτροπε, σας ζητώ να αποσύρετε την ΣΟΕΣ. Η συμφωνία αυτή με, την, με το μηχανισμό ISDS ε, αντιπροσωπεύει την ε, παράδοση της εθνικής κυριαρχίας της μεγάλης εταιρείας. Δεύτερον, η ΣΟΕΣ θα καταργήσει περισσότερες θέσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ότι αυτές που θα δημιουργήσουν οι πολυεθνικές για τις οποίες έχει ε, ε, σχεδιαστεί η ΣΟΕΣ. Επίσης, η συμφωνία αυτή θα καταστρέψει ε, τις μικρές ε, παραγωγές και τη μικρή κτηνοτροφία ε, βοήου κρέατος. όμως υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Έχουμε μιλήσει για την κλιματική αλλαγή σε αυτό το κοινοβούλιο το να αρχίσουν να κυκλοφορούν κάθε μέρα ε, ε, τρόφιμα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα μπορούσαμε να ε, παράγουμε και να καταναλώνουμε επιτόπου ε, αυτό αποτελεί, θα δημιουργήσει σημαντική, σημαντικό βάρος στο περιβάλλον με πολλές εκπομπές και προφανώς θα χειροτερεύσει την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαντρα Κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απασχόληση και η ανάπτυξη εξαρτώνται κυρίω από μια εμπορική πολιτική που θέλει να βοηθήσει τι επιχειρήσει και να εκμεταλλευτεί την ε, ε, ζήτηση. Γι' αυτό και ακριβώ είναι θεμελιώδη συμβασία σε αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να είναι προ όφελο διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και την αναγνώριση κάποιων γεωγραφικών ενδείξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εμπορικό εταίρος του Καναδά μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες και επομένως η συμφωνία αυτή είναι ζωτική σημασία, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα ISDS. Εάν αυτή η ρήτρα εφαρμοστεί, μια πολυεθνική που επενδύει σε μια χώρα θα μπορεί να προκαλέσει την κυβέρνηση μιας χώρας μέσω μιας διαδικασίας διεθνούς διαιτησίας ε, χάνοντας ουσιαστικά το εθνικό δικαστικό σύστημα και μπορεί να δημιουργηθεί μια παράλληλη δικαιοδοσία που δεν θα επιτρέπει στο κράτος να έχει τον τελευταίο λόγο για πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τίνει ευήκονους και να ακούσει τα όσα έχει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Καπούτο. Καθήκον βέβαια δεν είναι να ανακαλώ στην τάξη ενήλικες. Αλλά κύριε Καπούτο, μια και μόλις άρχισε η θητεία θα σας το επισημάνω, ξεκίνησε από την αρχή της παρέμβασης σας κύριε Καπούτο το κόκκινο φωτάκι που έχω εδώ μπροστά μου που σημαίνει ότι οι διερμηνείς σας καλούν να μιλήσετε πιο αργά γιατί δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Ούτε καν οι Ιταλοί ε, συμπολίτες σας θα μπορούσαν να σα παρακολουθήσουν πόσο δε μάλλον οι ε, ε, κάτοικοι οι Ευρωπαίοι όλη τη Υπήρου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν σα καλώ να φροντίσετε με με την ομιλία σας να βοηθήσετε και τους εξαίρετους διερμηνείς που έχουμε στη θέση μας να μεταφράζουν σωστά την ε, ομιλία σας. Σας ε, χτύψα το σφυράκι για να σας δώσω το ε, σημάδι ότι πρέπει να μιλήσετε πιο αργά. Εάν όμως συνεχίζετε θα είμαι υποχρεωμένος να αφήσω τους ερμηνείς να κλείσουν το μικρόφωνο, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάντι, παρακαλώ. Ε, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί, η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Ευρύτατη πρόσβαση στην αγορά για τι εισαγωγέ μα και τι εξαγωγέ μα και ε, σημαντική δυνατότητα για πλειοδοτικού διαγωνισμού και σε τοπικό επίπεδο. Και επίσης υπάρχουν και σημαντικές πρόοδοι στην προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων. Η πλειονότητα των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της διαπραγμάτευσης ε, αναγνωρίζονται πλήρως ε, στην αγορά της Βορειοαμερικής. Ε, περιοχή η οποία ήταν ε, εκτός ορίων για τον γεωργικό και διατροφικό μας τομέα. Είναι θετικό φυσικά το αποτέλεσμα, αλλά δεν μα ικανοποιεί απολύτω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στην προστασία των προϊόντων τη, ιδιαίτερα τα ποιοτικά τη προϊόντα παγκοσμίω. Και πέραν τη τεχνικής αξιολόγησης του κειμένου, η συμφωνία αυτή και η TTIP ε, στη συνέχεια είναι ιδιαίτερα σημαντικές, δεδομένου ότι εξελίσσονται οι σχέσεις ε, με συγκεκριμένο τρόπο με τη Ρωσία και με το τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλε διμερείς διαπραγματεύσει. Θα πρέπει σίγουρα να εμβαθύνουμε στον τρόπο επίλυση ε, διαφορών, το περιβόητο ISDS, και ε, επί τη βάση μιας συγκεκριμένη διαδικασίας διαβούλευσης. Θεωρώ ότι μια τέτοια ρήτρα δεν θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων εις βάρος ε, της αξιολόγησης αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Ντάντζ. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία Καρστιά και για να κλείσει η συζήτηση θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, σας πω για το ISDS, γιατί προφανώς ε, αυτό είναι το φλέγον θέμα για τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι περισσότεροι θα χάσουν τον ύπνο τους από όσους είναι παρόντες εδώ. θα απαντήσω λοιπόν σε άλλες ερωτήσεις. Αν και κύριε Λέχτριτ, εσείς νομίζω ότι μια χαρά θα κοιμηθείτε και το ελπίζω άλλωστε. Η πρώτη ερώτηση από τον κύριο Μάρτιν. Γιατί δεν ξεκινά ε, το Συμβούλιο, ε, δεν μονογράφει το Συμβούλιο αυτές τις συμφωνίες. Το Συμβούλιο δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο ποτέ στο παρελθόν. Η διαδικασία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία μονογράφει τις συμφωνία μετά από το νομικό έλεγχο και ο νομικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο Πρωθυπουργό ε, Χάρπερ ανακοίνωσαν στην ε, ε, Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει. Αυτό απαντά απλώ στην ερώτησή σα. Για τα γενώσιμα φάρμακα, βεβαίω μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Όχι μόνο με τον Καναδά, αλλά και με άλλες χώρες Για παράδειγμα, διαπραγματεύσει με την Ινδία, οι οποίε δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Και εκεί η προσέγγιση μας ήταν ότι δεν θα πρέπει να παρακολουθεί το εμπόριο σε γενώσιμα φάρμακα. Τα μη εμπορικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ε, τα TSN, θεωρήσαμε ότι αυτά ε, επαφίονται στον ΠΟΕ. Και αυτό ε, νομίζω ότι είναι δείγμα σοφροσύνης, αν και περιορισμένης. Όσον αφορά την εντολή και τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, θα επανέλθω στη δημόσια διαβούλευση, αλλά ως προς την εντολή θα πρέπει να διευκρινίσω ότι μας ζητήθηκε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για το ISDS. Αλλά θα επανέλθω στο σημείο αυτό αργότερα. Ο κύριος Μινέρ και κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν στη συμφωνία ως συμφωνία για τις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο και όχι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ξέρετε. Αυτές οι οποίες χρειάζονται συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι ε, αυτή η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα τους δώσει μια νέα αγορά και αυτό κάνουν αυτές οι συμφωνίες. Επομένως δεν ισχύει ο ισχυρισμός σας. Κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν στην πρόσβαση στη συμφωνία, ο κύριος Ζαντό, ο κύριος Λάγκε. Τα πράγματα είναι απλά. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, Απεστάλλει συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φαντάζομαι και σε εσά κύριε Λάγκε και στα κράτη-μέλη και το κείμενο της ΣΕΤΑ θα δημοσιευθεί αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ε, συντονίζουν τις θέσεις τους και ετοιμάζεται και μία εκδοχή για άτομα με προβλήματα όρασης ε, και φυσικά θα πρέπει να γίνουν και κάποιες ε, προσαρμογές και κατά πάσα πιθανότητα θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν κρατάμε τίποτα κρυφό, ξέρετε. Και δεν είμαι βέβαιος και ότι είναι τόσοι πολλοί πολίτες οι οποίοι είναι αναμονή της ε, ε, συμφωνίας για να τη διαβάσουν τα βράδια του φθινοπόρου. έχω τις αμφιβολίες μου. Έχω την αμφιβολία μου για το κατά πόσο θα τη διαβάσετε κι εσείς. ακόμα και αν ε, ε, αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση, είναι πολύ ανιαρά τα όσα θα διαβάσετε. Αυτό σε απάντηση και σε όσους φοβούνται ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι λέει το κείμενο. Κύριε Λεπέν, εξαφανίστηκε. Ήταν εδώ με πολλούς υποστηρικτές της, αλλά εξαϊλώθηκε μάλλον, δεν ξέρω τι κάνει. είπε ότι ελπίζει ότι για μια φορά θα ψηφίσετε σωστά. Κάθε φορά το ίδιο ζητάει, ξέρετε, και νομίζω ότι μάλλον δεν τη λαμβάνετε υπόψη σας. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να της εξηγήσετε γιατί. Κύριε Κέλλη, για το σύστημα των ποσοστώσεων, αλλά και ο κύριος Κέλλη εξαφανίστηκε. Φεύγουν όλοι εδώ, μου φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ε, μιλάω πολύ. Το σύστημα των ποσοστώσεων και τα ε, κρέατα καλής ποιότητας, ξέρετε ότι υπάρχει διαφορά ε, ε, πολύ σαφή ταξινόμηση και είναι πολύ σαφή η διαφορά μεταξύ των ε, κρέατων καλής ποιότητας και ε, των Δευτέρας Διαλογής και είναι πολύ ξεχωριστές οι αγορές και λαμβάνονται αυτά υπόψη. Υπήρχε και η ερώτηση της κυρίας Αρενά για το κατά πόσον θα αλλάξουμε τα πρότυπα για κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα, ε, σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ε, ε, κάτι τέτοιο προς συζήτηση. Τα πρότυπα αυτά τα έχετε καθορίσει εσείς κυρία Αρενά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Τώρα για τις πρωτοβουλίες των πολιτών, την ECI, Μία πρωτοβουλία πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να προτείνει κάποιο νομοθετικό κείμενο. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να προτείνει τη σύναψη μιας συμφωνίας με τρίτη χώρα. Αλλά δεν καλύπτει αιτήματα προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην κάνουν κάτι. Για παράδειγμα να σταματήσει η διαπραγμάτευση εμπορικής συμφωνίας όπως η TTIP ή να μην υπογραφεί μια συμφωνία όπως η ΣΥΤΑ. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί Από εκεί και πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αποφασίσουν. Επομένω, το αίτημα να μην ολοκληρωθεί η συμφωνία ΣΥΤΑ και να σταματήσουν οι διαπραγματεύσει για την TTIP θεωρούνται μη παραδεκτά αιτήματα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και ε, πολιτών και ε, επομένως ε, είναι πολύ, καθόλου ανώμημα τα κριτήρια. Μπορείτε κάλλιστα να υποβάλλετε ενστάσει και έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Τώρα, για το ISDS, το Σύστημα Επίλυσης Διαφορών Επενδυτών Κρατών. Ε, δεν ξέρω αν έχω ε, λίγο καιρό ε, επιπλέον κύριε Πρόεδρε γιατί τόσες πολλές ερωτήσεις ε, τέθησαν που σημαίνει ότι μάλλον έχετε χάσει τον ύπνο σας για το θέμα αυτό. Τον Απρίλιο του 2011 υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές πολιτικές επενδύσεων που εγκρίθηκε και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ε, στην οποία ε, υπερψήφισαν και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ζήτησε να υπάρχουν διαδικασίες ISDS, Ευρωπαϊκές Επενδυτικές Συμφωνίες, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία κατάχρηση του συστήματος. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο κίνησης της απάντησής μου. Το αυτό ισχύει και για την εντολή την οποία λάβαμε από το Συμβούλιο Υπουργών αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη εντολή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, ότι πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία, ε, μια ρήτρα ESDS ε στη συμφωνία. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά ξαφνικά αυτό έγινε το πλέον επίμαχο ζήτημα για τα θέματα εμπορίου. Και πολλά μέλη ανέφεραν τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. η οποία δείχνει ότι όλος ε, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, σκέφτεται ε, αντίστοιχα με αυτού. την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες εβδομάδες μάλλον, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της Δημόσιας διαβούλευση. Αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι υπάρχουν πάνω από 50.000 απαντήσεις από τις 150 περίπου χιλιάδες απαντήσεις που είναι ταυτόσιμες. Ε, συνήθως μπαίνει κάποιος ε, στην ιστοσελίδα, απαντάει στις ερωτήσεις και αποστέλει την απάντησή του. Ε, Κάποιοι απάντησαν ότι δεν γνωρίζω τίποτα, κάποιοι όμως ε, δεν καταλαβαίνουν τα τεχνικά, αλλά κατάφεραν ε, να στείλουν απάντηση χωρίς να κάνουν καμία εισαγωγή στο σύστημα και τελικώς έχουμε 50.000 ταυτόσιμες απαντήσεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε και 20.000 ταυτόσιμες απαντήσεις και υπάρχουν και καμιά 20.000 που λένε απλώς ότι είναι κατά. Θα τις δούμε όμως όλες τις απαντήσεις και αν υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία, σαφώς θα τα λάβουμε υπόψη. Τώρα, αν η ΣΥΤΑ αποτελεί προσχέδιο για την TTIP και άλλες αντίστοιχες συμφωνίες, ε, νομίζω ότι η ΣΥΤΑ, όπως και η συμφωνία με τη Σιγκαπούρη παρεμπιπτόντως, είναι σημείο καμπής για την αλλαγή προσέγγισης στις εμπορικές συμφωνίες και ε, ενισχύει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, ανανεώσει το σύστημα και θα σας δείξω και κάποιες καινοτομίες που έχουμε στη συμφωνία ΣΥΤΑ. Καταρχά υπάρχει ρητή αναφορά στη δυνατότητα κρατών να ε, νομοθετούν για το δημόσιο συμφέρον σαφής ορισμός ε, ε, προτύπων ε, προστασίας επενδύσεων για να μην υπάρχει Ε, Τρίτον, όλες οι ακροάσεις είναι δημόσιες, όλα τα έγγραφα είναι δημόσια για τους ενδιαφερομένους και παρεμπιπτόντως αυτά πηγαίνουν πολύ περαιτέρω από οποιαδήποτε διαδικασία σε εμπορικό δικαστήριο. Σε εμπορικό δικαστήριο το μόνο το οποίο είναι ανοιχτό είναι οι τελικές αποφάσεις. Δεν μπορεί κανείς να δει τους φακέλους των μερών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος νομικός εδώ, αλλά οι νομικοί το γνωρίζουν. Δεν μπορείτε να δείτε ε, τα στοιχεία του ε, αντισυμβαλόμενου. Ε, είναι πολύ πιο διάφανη λοιπόν η διαδικασία. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά δεσμευτικούς κανόνες ε, και υπάρχουν και εισαγωγή μιας αρχής η οποία επιτρέπει στους επενδυτές ε, να διαβεβαιώνει μάλλον ότι οι επενδυτές θα βαρύνονται με το κόστος ε, της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Και θα υπάρχει και κάποιος συγκεκριμένο φορέας ο οποίος θα βασίζεται στον αντίστοιχο φορέα του ΠΟΕ. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε συνέπεια στις αποφάσεις της διαιτησίας και οι διαιτητές θα είναι υπόλογοι και θα μπορούμε να προβλέψουμε και κάποια στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες βελτιώσεις στη Συμφωνία ΣΥΤΑ και ε, ίσως υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση στις επόμενες εμπορικές συμφωνίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι σαφές ότι η ΣΥΤΑ και η TTIP είναι δύο διαφορετικές συμφωνίες. Η ΣΥΤΑ έχει ήδη ε, συμφωνηθεί με τον Καναδά, έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαβίλευση, ενδιαφερόμενοι και οι πολίτες ε, ε μπορούν να δώσουν συγκεκριμένε απαντήσεις και ε, η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε στη διάρκεια της ε, διαβούλευσης ε, θα διαμορφώσει και τη θέση μας για την TTIP, ενώ η ΣΥΤΑ σε καμία περίπτωση δεν είναι προσχέδιο για την TTIP. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια πορεία η οποία είναι μονόδρομο. Σίγουρα δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε, αλλά τα όσα είχαμε βελτιωμένα στη ΣΥΤΑ θα βελτιωθούν περαιτέρω στι μελλοντικέ συμφωνίε. Ε, πολλά μέλη έθεσαν και το ερώτημα γιατί ε, χρειαζόμαστε στην στη ΣΥΤΑ δεδομένου ότι έχουμε ε, χώρες στις οποίες επικρατεί το κράτος δικαίου και έχουν συγκεκριμένα νομικά συστήματα. Πρέπει να έχουμε κάτι επιπλέον. Πρέπει οι Ευρωπαίοι επενδυτέ να μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζουν τα δικαιώματά του και γι' αυτό ακριβώ γιατί η συμφωνία ΣΥΤΑ δεν θα μπορεί να εφαρμόζεται στα δικαστήρια του Καναδά. θα είναι γιατί ε, είναι δυτή η προσέγγισή τους, ενώ εμάς είναι τελείως διαφορετική. Είτε είναι συμφωνία με τον Καναδά ή με τη Σιγκαπούρη, οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα ισχύει αμέσως από τα εγχώρια δικαστήρια, γιατί είναι ε, συγκεκριμένη η νομολογία στα ε, καναδικά δικαστήρια και δεν μπορούν να δώσουν σε εφαρμογή απευθεία συγκεκριμένε αποφάσει ε, σε διεθνέ επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν προστασία για του επενδυτέ. Η χάρτα ε, ενέργειας ισχύει για πολλά κράτη-μέλη ήδη και ακόμα και τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουν αρκετές ε, επενδυτικέ συμφωνίε μεταξύ τους. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, από τις 271 ε, υποθέσεις που έχουν καταγραφεί από το 2007 μέχρι το 2013, το, 50, το 15%, 40 ε, περίπου δηλαδή υποθέσεις, είναι ενδοκοινοτικές υποθέσεις. Υποθέσεις οι οποίες ξεκίνησαν από επενδυτές από ένα κράτος μέλος κατά κάποιο άλλο κράτος μέλος. Και εμείς παρεπιπτόντως έχουμε προτείνει ότι θα υπάρχει και κάποιος επιπλέον κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά κράτη-μέλη και το δικό σας το κράτος μέλος αρνήθηκαν. Κύριε Ελένε. Να υπάρχει επιπλέον ρήτρα για ε, συμφωνίες με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην ε, πολιτική που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν συμφωνίε με τον Καναδά και άρα μόνο οι δικοί του επενδυτέ είναι προστατευμένοι στον Καναδά, ενώ των άλλων κρατών οι επενδυτέ όχι. Εν τέλει, είναι ένας τρόπος να εισαχθεί ένα σύστημα, να εισαχθούν αλλαγέ στο σύστημα ISDS και να αποτελέσει έτσι ένα πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα. Θυμάμαι πολύ καλά ότι είχε γίνει μια δημόσια συζήτηση στο Βερολίνο με συμμετοχή του Μάικ Φόρμαν και του υποφαινομένου του κυρίου Σίγμαρ Κάμπριελ, αντιπρόεδρο της κυβερνήσεώς σας και μια συζήτηση από τις πολύ ζωντανές, από αυτές που μου αρέσουν πολύ, που σε τελευταία ανάλυση γι' αυτό έκανα πολιτική 40 χρόνια τώρα, ε, και είπε στο τέλος ο κύριος Ζίγμαρ Κάμπριελ ότι ε, υπάρχουν και θετικά στοιχεία, παραδείγματα είναι πολύ δύσκολο να απορριφθεί η ISDS με τις ΗΠΑ ή με τον Καναδά και να ζητούμε να γίνεται μια ISDS σε σχέση με την Κίνα, ένα ε, μηχανισμό επίλυση διαφορών. Άρα λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε πρότυπα τα οποία θα μπορούμε να διαδώσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό πιστεύω να το αντιληφθεί το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Μίλησατε περισσότερο από ό,τι υπολόγιζα. Αλλά μια και χθε το βράδυ μίλησατε πολύ πιο σύντομα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Σας επέτρεψα να μιλήσετε. Ε, θα παρακαλέσω όμως ε, στο μέλλον να απαντάτε για τους βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται στο ημικύκλιο, γιατί βέβαια δεν είναι σωστό κάποιο να διατυπώνει ερωτήσει και να αποχωρεί. Κλείνει λοιπόν εδώ η συζήτηση για το θέμα αυτό και περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη που είναι δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωέ στην Ευρώπη. Και εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει το λόγο η Επίτροπο Χέντιγκορτ. Περιμένουμε μερικά λεπτά μόνο. Κύριε Λάιχτφριτ, εσεί θα συνοδεύσετε τον Επίτροπο που αποχωρεί και μπορεί να ξεκινήσει η κυρία Χέντιγκαρτ.